Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε πολλά θέματα. Καλωσορίζω τους παρόντες. Οπότε, ε, αν αρχίσουμε με την ημερήσια διάταξη προχθές, ο πρόεδρος Σούλτς με ενημέρωσε ότι η ομάδα εργασίας, η ομάδα επαφής για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου συμμετέχω ε, θα γίνει σήμερα είναι η σχέση μεταξύ του πολιετούς πλαισίου και της συναπόφασης οπότε πρέπει να συμμετάσχω προτείνω λοιπόν να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη οι ψηφοφορίες να πάνε στις 11 γιατί πρέπει να συμμετάσχω στη συνεδρίαση της ομάδας επαφής εάν συμφωνείτε παρακαλώ και τους συνεργάτες των ε, συναδέλφων βουλευτών να τους ενημερώσουν θα συζητηθούν πριν άρα θα συζητήσουμε το 14 του κυρίου Σταυρακάκη και ενδεχομένως αν έχουμε χρόνο και την γνωμοδότηση του κυρίου Ντόιτς για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά αμέσως μετά την έκθεση Βλάσακ. Ε, δεν βλέπω αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις αλλαγής της τη διάταξης. Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανή από το ίντερνετ. Βεβαίως οι χρόνοι είναι πάντα ενδεικτικοί, γιατί μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτα. Περνάμε στο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 29 και 30 Μαΐου. Τα πρακτικά έχουν διανεμηθεί. Θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν στο τέλος της συνεδρίασης εάν δεν έχουν υποβληθεί τροποποιήσεις. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Μόλις ενημερωθήκαμε, και αυτό ίσως είναι πρόβλημα, ότι η γνωμοδότηση που αποφασίσαμε να κάνουμε για τον ε, οριζόντιο κανονισμό της άμεσης πληρωμές και την ανάπτυξη της υπαίθρου είχαμε συμφωνήσει να γίνει από τον κύριο Κούρσκι. Όμως η γραμματεία της Άγκρη μας ενημέρωσε επειδή είναι πήγον ότι αποφάσισαν να ψηφίσουν την έκθεση στις 8 Ιουλίου, άρα ήδη την ψήφισαν και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 3 Σεπτεμβρίου και η έγκριση της έκθεσης στην Άγκρη θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. Άρα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ακόμη και την ταχύτερη συνήθη διαδικασία για τη γνωμοδότησή μας αυτή. Οπότε παρακαλώ όσοι επιθυμούν να υποβάλουν μεμονωμένα απευθείας στην άγκρη. Έχετε σχόλια από αυτού παρακαλώ. Όχι. Να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Είναι έκθεση του κ. Ότζικ Βλά... Θα πρέπει να αποφασίσουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών αλλά να αρχίσουμε με την παρουσίαση της έκθεσης από τον Ότζι και μετά θα έχουμε τα σχόλια των ε, ε σχεδόν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας ζητήσω να φορέσετε τα ακουστικά σας, γιατί θα ήθελα να μιλήσω στα τσεχικά, την μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Επιτρέψτε μου να πω ευθύ εξ αρχή ότι καλωσορίζω την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους που διαθέτουμε. Φροντίσαμε το θέμα να το καλύψουμε σε δύο τμήματα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να υπάρξει συστηματοποίηση και συστηματική χρήση της αρχής απλούστευσης. Γι' αυτό στο πρώτο μέρος αυτής της έκθεσης ασχολούμαστε με την διαδικασία top-up, ε, δηλαδή της ανάντι προσπάθειας μέχρι το 2013 και ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό από το 2014 έως το 2020. Ο κανονισμός ως τώρα έχει αποδείξει ότι είναι καλός και μπορεί να λειτουργήσει και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την άλλη, είμαι υπέρ της συστηματοποίησης και του δεύτερου σκέλους αυτής της έκθεσης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κανόνας 1 3 μπορεί να παραταθεί με την εξαίρεση των κρατών συνοχής για το 2007-2010 υπέρ του 1 συν 3 τάσουμε λοιπόν υπέρ του 1 συν 3 μεταξύ του 2013-2020 ο κανόνας αυτός έχει αποδείξει ως τώρα ότι είναι αποτελεσματικός επί μία διετία δεν εφαρμόστηκε Οπότε θεωρούμε ότι μπορεί να επανεισαχθεί. Υπάρχουν κονδύλια στον προπολογισμό, δεν ζητούμε κάτι επιπλέον για αυτό το μέτρο και απλώς να σας πω ποια είναι η συλλογιστική μας. Ότι πρώτα απ' όλα θα βασιζόμαστε στους στόχους και θα πρέπει η πολιτική συνοχής να ενισχύσει τις χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα. Ο κανόνας εν συν 3 θα πρέπει να διατεθεί και να ισχύει για τις χώρες που χρειάζονται περισσότερη ευελιξία. Επίσης, στόχος θα πρέπει να είναι χώρες οι οποίες έχουν πρέπει μάλλον να ευθυγραμμίσουν, να εξορθολογήσουν τον προπολογισμό τους, να υποβάλουν τα προγράμματα προσαρμογής τους ή να πραγματοποιήσουν αποταμιεύσεις για την περίοδο 2013-2020. Το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν, που ξέρουμε ότι δίνουν αποτελέσματα, και να υπάρξει μια κατάλληλη μετάβαση από το διάστημα αυτό στην επόμενη περίοδο. Οι χώρες αυτές, οι χώρες που αφορούν που αφορά αυτός ο κανόνας, δεν θα πιεστούν να διαλέγουν προγράμματα εάν δεν τα θεωρούν κατάλληλα. Και τέλος, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου όλοι προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να ενεργοποιηθούν νέοι μηχανισμοί και αυτές οι χώρες να έχουν περισσότερους πόρους, περισσότερα κονδύλια στη διάθεσή τους. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Αλλά ούτε και υπάρχει χρόνο, ε, ούτε υπάρχει λόγο μάλλον να μην δοθεί χρόνο στι χώρε αυτέ εφόσον το χρειάζονται. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι είναι απαραίτητο, εφόσον υπάρχουν τα κονδύλια, να βρούμε και μηχανισμού για να διατίθενται αυτά. Επίση, δεν θέλουμε να γίνουν όλε οι προσπάθειε αποταμίευση ή εξοικονόμηση στο τέλο τη περίοδου, περίοδου προγραμματισμού. στόχος είναι να δώσουμε σε αυτές τις χώρες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα σταδιακά και να υποφεληθούν από αυτά σταδιακά. Δεν χρειάζεται να κοινοποιούνται όλα σε κάθε χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρχει επαρκή ευελιξία για να κάνει η Επιτροπή αυτό που θεωρεί το καλύτερο για την κάθε περίπτωση. Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή από πλευρά μου και δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις παρεκκλήσεις και τις εξαιρέσεις της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, όπως τώρα ισχύουν, η δική μου λύση είναι να δούμε τι ενδεχόμενα προβλήματα μπορεί να υπάρξουν με άλλες χώρες που ίσως αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντόιτς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όσα είπε ο κύριος Βλάσακ είναι ορθά. Εξάλλου πάντα είναι σύντομος, κάτι το οποίο εκτιμώ όλος ιδιαίτερος, παρόλο που το θέμα είναι σημαντικό πάντα. Είναι πολύ λογικός λοιπόν ο σύντομο και έτσι θα προσπαθήσω και εγώ να ακολουθήσω το παράδειγμά του. Έχω να σας αναφέρω τέσσερα θέματα σχετικά με το θέμα αυτό. Εκ μέρους της δικιάς μου πολιτικής ομάδας βέβαια. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον κύριο και για το έργο του. Πιστεύω ότι το κείμενο αυτό περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά ζητήματα και εγώ προσωπικά και η πολιτική μου ομάδα συμφωνούμε με το κείμενό του. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξή. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει απώλεια ή κίνδυνος απώλειας πόρων. Και πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι για απώλεια πόρων. Εάν αυτή η αυτόματη απώλεια λάβει χώρα, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο πρόκειται για μια ορθή απόφαση ή όχι. Όσον αφορά τώρα τα κονδύλια συνοχής, υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα για τις διάφορες χώρες και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι αποδέσμευση τελικά πρέπει να αναμένουμε. Όλα αυτά τα κονδύλια λοιπόν που έχουν να κάνουν ε, με την κάθε χώρα χωριστά θα πρέπει κάθε χώρα να μπορεί να ε, τα χρησιμοποιεί όσο γίνεται καλύτερα. Πιστεύω συνεπώς ότι οι χώρες μέλη καμιά φορά κάνουν λάθη, έχουν προβλήματα στην εκτέλεση των προγραμμάτων. Είναι αλήθεια, υπάρχουν τα προγράμματα και τα προγράμματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια πόρων. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό και δεν είναι μόνο η κρίση. Υπάρχει κρίση βέβαια που είναι εδώ από το 2008-2009, μια κρίση η οποία σίγουρα είναι υπεύθυνη για πολλά προβλήματα, γιατί η κρίση είναι αυτή που δυσκόλεψε τόσο πολύ την εκτέλεση των προγραμμάτων. Δεν το περιμέναμε, δεν μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει αυτή την κρίση. Οπότε, ε, καταρχήν, η κρίση είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι πολλές χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια έχω μια τροπολογία σχετικά με τη Σλοβακία και την Ρουμανία. Πιστεύω ότι ο κίνδυνος υπάρχει όχι μόνο για τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, αλλά και για άλλες χώρες. Αυτό λέει η τροπολογία μου. Έπειτα, όσον αφορά τον κανόνα νη συν 3, συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Βλάσεκ. Και πιστεύω ότι Όλα αυτά θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα στο κείμενο με τη βοήθεια μιας τροπολογίας για να αναφερθούμε στο έτος 2013 και για να πούμε ότι τα λογιστικά πρέπει να είναι έτοιμα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Όσον αφορά το top-up, για την ε, ονομασία που έχει να κάνει με τον κανονισμό για το top-up, νομίζω ότι εδώ πρέπει να αλλάξει κάπως το κείμενο για το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Πρόκειται για μια αύξηση 10% στην συγχρηματοδότηση. Και είναι κάτι που πρέπει να αφορά όλες τις χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και που δεν είναι πια χώρες μέσα σε πρόγραμμα, που δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να έχουν κανονικά αυτή τη βοήθεια. Πρόκειται για χώρες οι οποίες δεν είναι πια σε πρόγραμμα ε, δημοσιονομικής εξυγένσης, αλλά συνεχίζουν να έχουν ανάγκη από βοήθεια. Χρειάζονται δηλαδή τη βοήθεια αυτή για να μπορέσουν να ε, πληρώσουν ε, τα έξοδα. Σε αυτή τη μεταβατική λοιπόν περίοδο η αύξηση της χρηματοδότησης πρέπει να αφορά και αυτές τις χώρες. Με τις τροπολογίες αυτές λοιπόν μπορώ να στηρίξω απόλυτα το κείμενο του κύριου Βλάσακ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαστινάρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βλάσα για την έκθεσή του. Όπως είπα και την τελευταία φορά, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, η πρόταση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τεράστια σημασία γιατί ο στόχος της είναι να βοηθήσει χώρες οι οποίες για έναν ή τον άλλο λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα ή κινδύνους και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν την ιδέα που βρίσκεται πίσω από την πρότασή του, ιδιαίτερα όταν προτείνει να γενικευτεί η πρόταση αυτή για την Σλοβακία και τη Ρουμανία και όταν προτείνει επίσης και κάποιες άλλες αλλαγές για να βοηθήσει χώρες δηλαδή η γενίκευση του κανόνα νήσιν 3. Όμως πρέπει να μην ξεχνάμε τι βρίσκεται πίσω από την πρόταση αυτή, ποιο είναι το πλαίσιο και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση. Ένας λόγος είναι ότι πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ή μέσα σε προγράμματα δημοσιονομικής εξυγένσης. Ένας άλλος λόγος όμως είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όσα έχουν αποφασίσει ομόφανα όλοι οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων τη νύχτα εκείνη της 8 η Φεβρουαρίου. Κάτι στο οποίο συμφώνησαν και 27 χώρες μέλη. Δεν ήταν δηλαδή κάτι μόνο για Ρουμανία και Σλοβακία. Όλοι συμφώνησαν στον κανόνα αυτό. Συνεπώς, πρέπει να θυμόμαστε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Συμβούλιο. Ότι να δούμε δηλαδή κατά πόσο υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν αν υπάρξει απόκληση από τη συμφωνία αυτή του Φεβρουαρίου. αν δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε τη συμφωνία. Δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση. Και ξέρουμε ήδη πόσο δύσκολο ήταν πριν από δύο εβδομάδες να επιτευχθεί νέα συμφωνία με το Συμβούλιο μετά από την απειλή του Κοινοβουλίου σε πιο ψηλό επίπεδο. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Να ξέρουμε ότι ο χρόνος περνάει και ο χρόνος δεν είναι εχθρό μόνο για τι δύο αυτέ χώρε, αλλά και για ολόκληρο το Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει έγκαιρα να εγκρίνει του γενικού κανονισμού και του ειδικού κανονισμού. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αν δεν υιοθετήσουμε έγκαιρα αυτή ή κάποια άλλη λύση, τότε θα είναι άχρηστο. Γιατί πρόκειται για το 2011 και το 2012 και με την εφαρμογή του κανόνα νη συν 3, εάν χάσουμε και το 2013 και δεν εγκρίνουμε έγκαιρα τη λύση, τότε η λύση δεν θα έχει πια νόημα. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να γίνει γρήγορα. Άρα θα έλεγα να μην αλλάξουμε την πρόταση της Επιτροπής και να φροντίσουμε να την εγκρίνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τότε θα έχουμε αρκετό χρόνο ώστε να πετύχουμε την τελική συμφωνία και την καλή εφαρμογή. Διότι το θέμα δεν είναι να δείξουμε ε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε απέναντι στη μία την άλλη χώρα. Εντάξει, ευχαρίστως, θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τροπολογίες για να έχουμε τη συμφωνία σε δύο στάδια. Πρώτα για τη Σλοβακία και τη Ρουμανία να βασιστούμε στην πρόταση Επιτροπής χωρίς αλλαγή και μετά να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο βήμα για άλλες χώρες οι οποίες θα θέλανε να χρησιμοποιήσουν την ίδια ρύθμιση. Αλλά για αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει πρώτα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Σημαίνει ότι θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώ αυτή θα είναι η δικιά μου τροπολογία για μία λύση σε δύο βήματα. Πρώτα Ρουμανία-Σλοβακία και μετά για τις υπόλοιπε χώρες ενδεχομένω, και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Και αυτή είναι η έκκληση που κάνω σε όλους σας. Προσπαθήστε να με καταλάβετε και το τελευταίο που θέλω να σας πω. Μετά από τις φοβερές προσπάθειες που έχει κάνει η ρουμανική κυβέρνηση έχουμε τριπλασιάσει την απορρόφηση των κονδυλίων σε σχέση με το 2012. Παρόλα αυτά εξακολουθούμε να είμαστε σε επίπεδο 19% απορρόφησης πληρωμών, έτσι. Αν τώρα δεν πάρουμε την απόφαση και όχι Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημέρωση που μας έκανες και αυτό το χαρτί που μας έδωσες. Η Ρουμανία, βάσει των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κινδυνεύει να απολέσει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό. Συνεπώς, σας ξαναλέω, λάβετε υπόψη σας αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει ευελιξία. Δεν ε, κάνει διάκριση σε βάρος κανενός, Ας κάνουμε αυτό που είναι εύκολο να πετύχουμε τώρα γρήγορα με τη Σλοβακία και τη Ρουβανία και μετά ας περάσουμε στο δεύτερο βήμα Α είναι αυτό ο συμβασμό για να δούμε αργότερα τι θα γίνει με τι υπόλοιπε χώρε. Και μην ξεχνάτε για το εξή, κυρία Πρόεδρε. Η εφαρμογή του κανόνα νη συν 3 και η γενίκευση του κανόνα αυτού για το 2014 μέχρι το 2020 σημαίνει ότι ξαναρχίζει ο τριμερής διάλογος, γιατί έχουμε τον γενικό κανονισμό που έχουμε ήδη διαπραγματευτεί, το ξέρουν οι συνάδελφοι. Δεν Βλέπω η Κωνσταντσα Κρέλ και ο κύριος Φανίστεροι. Ε, δεν ξέρω αν θέλουν να ξαναρχίσουν νέο τριμερή διάλογο για τον κανόνα νήσιν 3 για την ε, ε, πολιτική συνοχή. Φαντάζομαι πως όχι. Ευχαριστώ. But, Ναι. Δεν βλέπω τον κύριο Χρυσόγελο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους πράσινους να πάρει το λόγο. Όχι, περνάμε στον κύριο Νικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σλοβακικά. Και πρέπει να πω ότι κοιτάζοντας τις αδρές γραμμές της πρότασης, δύο σχόλια πρέπει να κάνω ότι εκτιμώ την οπτική γωνία του κυρίου Βλάσακ και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένας γνώστης του αντικειμένου. Έχει μελετήσει βαθιά το θέμα. Να επισημάνω κάποια στοιχεία τα οποία εφόσον ληφθούν υπόψη θα επιτρέψουν να η πρόταση και να αποτελεί ένα πραγματικό βήμα πρόοδου αλλά να αντικατοπτρίζει και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ως τώρα μετά τους ε, προηγούμενους ομιλητές και όπως είπαν και εκείνοι θα πρέπει να μην ξεχνάμε τι συνέβη και στο Συμβούλιο με τη συμφωνία μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων υπήρξαν χώρες που υπέβαλαν συγκεκριμένα αιτήματα λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζουν και χώρες γειτονικές της Σλοβακίας μέσω των διαπραγματεύσεων, συγκεκριμένα η δημοκρατία της Τσεχίας, απέσπασε 900 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλω να περάσω όμως σε λεπτομέρειες. Η Σλοβακία και η Ρουμανία ακόμη χρηματοδοτούνται με κάποια κονδύλια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να απορροφηθούν. Γι' αυτό ζητούμε να εισαχθεί μια αρχή που θα επιτρέπει την απορρόφηση των προβλεπόμενων κονδυλίων, τα οποία όμως ακόμη δεν έχουν εκτεμευτεί. Έτσι έχει τοποθετηθεί η Σλοβακία στο Συμβούλιο. Και για αυτά που είπε ο κύριος Βλάσακ, δεν θα πετήσουμε δεν θα ζητήσουμε περισσότερους πόρους. Απλώς θα θέλαμε να μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο να απορροφήσουμε τα κονδύλια που προβλέπει η πολιτική συνοχής. Θέλουμε λοιπόν να έχει γενική ισχύ αυτή η αρχή. Και εδώ πρέπει να ε, συμφωνήσω με την πολύ πραγματιστική προσέγγιση του εισηγητή και το διαχωρισμό της ε, περίπτωσης αυτής σε δύο σκέλη. Σε μία πρώτη φάση μπορούμε να εγκρίνουμε τον καρονα αποδέσμευση συν 3 για τη Σλοβακία και τη Ρουμανία και σε μια δεύτερη φάση θα μπορούσαμε να δούμε πώς η αρχή αυτή ενδεχομένως να επεκταθεί και να ισχύσει και για άλλες χώρες. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα διτράξουμε την ισορροπία που έχει επιτευχθεί μέχρι των διαπραγματεύσεων και θα συμφωνούμε και με την αρχή που έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη θαυμάσια εργασία, πραγματικά εργασία υψηλού επίπεδου του συναδέλφου μου κυρίου Βλάσσα. Όλα όσα υπόθηκαν από αυτού είναι σωστά, κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Όμως, αυτό που μας προτείνει ο κύριος Βλάσσακ, δηλαδή μια λύση συστημική, θα επιτρέψει σε ορισμένες χώρες να απορροφούν πόρους και φυσικά πρέπει να λάβουμε τα προβλήματα της Σλοβακίας και της Ρουμανίας αλλά τόσο γενικότερη θα ήμουν λοιπόν υπέρ του να προστατεύσουμε τη Ρουμανία και τη Σλοβακία αλλά να το επεκτείνουμε σε όλες τις χώρες είναι συζητήσιμο. Όχι, είναι συζητήσιμο, αλλιώς αργότερα να χρειαστεί να το ξαναδούμε, τώρα να το εφαρμόσουμε για όλες τις χώρες, συμφωνώ. Να αναφέρω όμως κάτι που μπορεί να μην το αντιλαμβανόμεθα από πρώτη άποψη, αλλά όντως άμα το σκεφτούμε επηρεάζει την κατάσταση στα κράτη-μέλη όταν ε, εκπονούν προγράμματα, ζητάνε ε, πληρωμές κτλ. Ξέρετε ότι σε κάποιες χώρες συνοχής υπήρξαν ε, πολύ σοβαρές πλημμύρες. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να κάνουμε έκκληση στην Επιτροπή να το λάβει υπόψη. Πρέπει να λεφθεί υπόψη αυτή η επιβαρυντική κατάσταση, δηλαδή τουλάχιστον να μην απαιτηθούν ε, αυστηρές προδιαγραφές ή να μην ερμηνευτούν αυστηρά οι κανόνες ε, λόγω των προβλημάτων ε, που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές. Όπως είπα, οι συστημικές λύσεις είναι οι καλύτερες. Αλλά παρόλα αυτά μάλλον τίνουμε προς μια πραγματιστική λύση με έναν κανονισμό για την Ρουμανία και την ε, Σλοβακία και η συστημική λύση σε μεταγενέστερο σχέδιο ευχαριστώ. Σε μεταγενέστερη φάση ευχαριστώ. Ο Βλάντιμιρ Μάνκ. Ευχα... Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο και για τις ε, πολύ ρεαλιστικές του προτάσεις και τις προτινόμενες λύσεις. Είναι πραγματικά η σωστή τοποθέτηση αυτή που προτείνει, γιατί ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι έχει τεχνογνωσία στον τομέα αυτό. Τώρα για τις διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα είναι να διατηρήσουμε την ισορροπία στην οποία καταλήξαμε και να έχουμε υπόψη και τις εξελίξεις στον κανονισμό για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι εναλλακτικέ που προτείνει ο κύριος Βλάσακ, εφόσον εγκριθούν από το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο, τότε θα μας ε, επιτρέψουν να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, που όμως έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμφωνήσει. Θα καταρρεύσουν τα πάντα αν δεν υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Γι' αυτό το λόγο, ίσως η καλύτερη λύση να είναι να εγκρίνουμε την πρόταση του Συμβουλίου, τέλο πάντων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ίσω σήμερα κιόλα. Θα μπορούσε μάλιστα να διαιρεθεί η έκθεση του κυρίου Βλάσακ σε δύο τμήματα. Η μία να παρουσιαστεί ω πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλη ω πρόταση του κυρίου Βλάσακ. Α κάνουμε κι εμεί μια παραχώρηση, μια προσπάθεια για να προχωρήσουμε και να προχωρήσει το όλο θέμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ματούλα. Ματούλα. Και εγώ να συγχαρώ τον ε, κύριο Βλάσσα για την έκθεσή του η οποία ε, παρουσιάζει αναλυτικά τα κράτη-μέλη που έχουν ε, επηρεαστεί ή αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές κατά της χρηματοπιστωτικής τους σταθερότητας. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να επιδιώξουμε να επιτύχουμε τους στόχους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να τροποποιήσουμε το κανονισμό 1083 λόγω της ε, οικονομικής κρίσης και η συμφωνία στο Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου και τα πορίσματα επίσης πρέπει να λεφθούν υπόψη. Η πρόταση της Κομισιόν επιδιώκει μια λύση ούτως ώστε δύο κράτη-μέλη, η Ρουμανία και η Σλοβακία, να λάβουν ε, εξαίρεση ε, στα πλαίσια του 1 συν 3 ούτως ώστε ε, οι κανόνες αποδέσμευσης να βασιστούν σε αυτό το 1 3 για το 2012. Όπως έχει υποβληθεί η πρόταση της Κομισιόν, θέλει να παραταθεί η περίοδος πριν υπάρξει αποδέσμευση για την Ρουμανία και τη Σλοβακία και δεύτερον, η πρόταση της Επιτροπής είναι απόλυτα λογική και βασίζεται σε ομόφανη ε, πρόταση στο Συμβούλιο. και προσπαθεί ε, να αντιμετωπίσει το διπλό ε, ανώτατο όριο για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Φυσικά υπάρχει θέμα ε, μεταφοράς υπάρχει θέμα αύξησης χρηματοδότησης κατά 10%. Αυτό ενδιαφέρει όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά που είπε ο κ. Μποστινάρου απλοποιούν και για μένα την επιχειρηματολογία. Πρέπει να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο. Και τονίζω ότι το Φεβρουάριο υπήρξε συμφωνία στο Συμβούλιο για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Υπήρξαν ε, επίσης άλλες ρυθμίσεις για άλλα κράτη-μέλη και νομίζω τώρα ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει υπερβληθεί το αδιέξοδο και θα συμβάλλουμε και εμείς αυτό εγκρίνοντας την πρόταση της Επιτροπής και νομίζω ότι θα χρειαστεί να υποστηρίξουμε και άλλα κράτη-μέλη στο μέλλον. Επ' αυτό ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανίστελρο. Ευχαριστώ, πολύ. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά αυτή που έχετε κάνει. Πρέπει να δούμε βέβαια όλες τις δυνατότητες και τελικά να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο βέβαια θα εγκριθεί. Οπότε παρακολουθώ τη συζήτηση και είναι σαφές ότι πρέπει να επιτελέσουμε το νομικό έργο. Σε αυτό το στάδιο δηλαδή πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Και πρέπει να πούμε ναι. Εγώ λέω στο διακανονισμό αυτό για τις δύο χώρες. Και μετά δεν βάζουμε κόμμα, βάζουμε ανωτελεία και μετά ζητάμε δύο πράγματα, ό,τι θέλουμε σε κάποιο άλλο στάδιο. Γρήγορα, μπορούμε να το ζητήσουμε, δεν θα είναι όμως γρήγορα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαπραγμάτευση για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχα έξι από τις χώρες του Βίζιγκράτ οι οποίοι ήρθαν και μου ζήτησαν ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Πολύ ωραία συζήτηση αυτή, αλλά δεν θα υπάρξει στήριξη στο Κοινοβούλιο. Ούτε από το ΕΛΚ, δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες. Πάντως πρέπει να πούμε ναι σε αυτό το στάδιο. Τελεία. Και μετά να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλουμε, αλλά σε αυτό το στάδιο πρέπει να πούμε ναι σε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι το πολιτικό μου μήνυμα και αυτό θέλει να περάσει και το ΕΛΚ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Μόνικα Σμόλκοβα τώρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η προλαλή σας με κάλυψε απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και με αυτό που είπε ο κύριος Μποστινάρο. Αυτό θα ήθελα και εγώ να εκφράσω. Είπε ο κύριος Μποστινάρο ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται και όχι εκτός και μας παρουσίασε το πλαίσιο. Οπότε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των κυρίων Τόιτσε και Λάσακ στα σημεία 50, 51 και 52 των αποφάσεων του Συμβουλίου, όπου αναφέρονται σε άλλες διατάξεις για ειδικά κονδύλια. Ο κίνδυνος είναι ότι αν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα νη 3 σε όλες τις χώρες και αποτύχουμε η Ουγγαρία ίσως τότε να χάσει επιπλέον κονδύλια της τάξεως του 1,56 δισεκατομμύρια ενώ προσπαθούν να πετύχουν 695 εκατομμύρια και δυνεύουν να χάσουν σε αυτή την περίπτωση 1,56 δις. Η Τσεχία που θα έπαιρνε 100 εκατομμύρια, τώρα κινδυνεύει να χάσει 530. Συνεπώς, πρέπει να δούμε τι έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Η Σλοβακία και η Ρουμανία δεν ζητούν επιπλέον κονδύλια. 21 χώρες ζητούν επιπλέον κονδύλια όμως. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο σύνολό τους. σε σχέση με τα επιπλέον κονδύλια για άλλες χώρες που θέλουμε να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Αν είχαμε άλλον ένα χρόνο, τότε ναι, θα θέλαμε ο κανόνας νη συν να γενικευθεί για την επόμενη χρονιά. Όμως δεν έχουμε χρόνο, οπότε ας εγκρίνουμε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε και μετά να δούμε πώς θα ζητήσουμε τα επιπλέον κονδύλια. Πρόεδρος, δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους στον κατάλογο μιλητών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο Ανδρέας Φανμπούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί έχουν επιλεγεί αυτές οι δύο χώρες. Ευχαριστώ. Η πρότασή μας βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα πορίσματα για το πολιετές πλαίσιο και βασισμένη σε αυτά τα πορίσματα προβλέψαμε λοιπόν εξαίρεση για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Γιατί μόνο για αυτές τις δύο, γιατί τα πορίσματα βασίζονται στον ε, δημοσιονομικό συμβιβασμό βασίζονται στο επίπεδο πόρων λοιπόν του προπολογισμού, οπότε προβλέφθηκε σημαντική μείωση του ΡΑΛ και αν ε, εφαρμόζαμε το 1 3 για όλες τις χώρες θα υπήρχε ε, ε, σημαντική δημοσιονομική επίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν επεκτάθηκε το, η δυνατότητα να αποφευχθεί η αποδέσμευση στη βάση του δημοσιονομικού συμβιβασμού που είχε συμφωνηθεί και με το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν εμένει στη θέση της για τον κανόνα 1-2, 1-3 όπως προτείνεται στην πρόταση. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτές τις διατάξεις. Βεβαίως, για την περίοδο 14-20 προβλέπεται το 1-3 για όλες τις χώρες, αλλά αυτό θα βασιστεί σε ένα νέο συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίσαμε για να εφαρμόσουμε στο μέλλον. Προσπαθούμε δηλαδή να απλοποιήσουμε και δεν θα διατηρήσουμε λοιπόν εξαιρέσεις. Για το δεύτερο σημείο, δηλαδή η παράταση του top-up της αύξησης της χρηματοδότησης των χωρών που θα είναι στον ε, μηχανισμό δημοσιονομικής στήριξης μετά το 2013 Η Επιτροπή μελέτησε τις διάφορες προτάσεις και τις συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο και θεωρεί όπως και ο κύριος Ντόιτς ότι ίσως θα ήταν σκόπιμο και εποφελές να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης μετά την έγκριση του CPR μετά για την επόμενη περίοδο. Θα μπορούσε λοιπόν η Κομισιόν να αποδεχθεί αυτήν την πρόταση. Αλλά πρέπει βέβαια να εγκριθεί συνολικά και να το εναρμονίσει με τις συζητήσεις για το CPR δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2016 Οπότε θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το το ακόμη τότε. Να δούμε πόσο θα διατηρηθεί αυτή η επέκτασή του. Τώρα για την ε, ευελιξία. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής είναι κατά της ευελιξίας γιατί οι χώρες μέλη μπορούν να ζητήσουν να αλλάξουν τα προγράμματα μέχρι το τέλος της περίοδου επιλεξιμότητας, δηλαδή στο τέλος του 2015. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις Επιτροπές Εποπτείας, δηλαδή τους εμπλεκόμενους φορείς ε, στα προγράμματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αποφασίσουν εάν χρειάζονται τροποποίηση. Αυτή η ευελιξία του 10% πρέπει βεβαίως να ε, είναι διαφανής, να μπορούν και οι υπηρεσίες της Κομισιόν και όλοι οι άλλοι φορείς να μελετήσουν πώς, τι αποτελέσματα έχει αυτή η ευελιξία. Αλλά θα πρέπει αυτή η ευελιξία να αφορά ε, ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, 10% σε... Γι' αυτό είναι σημαντικό επειδή θα υπάρχει τόσο μεγάλη επίπτωση σε σχέση με την αρχική απόφαση, να μελετήσουμε αν είναι σκόπιμο τόσο μεγάλο ποσοστό για την ευελιξία. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις, υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 17 Ιουλίου, 12 ώρα το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε, προβλέπουμε, στην συνεδρίασή μας το Σεπτέμβριο, δηλαδή στις 23 Σεπτεμβρίου, ούτω ώστε να περάσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, για να το κλείσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Σαβρακάκη να συζητήσει. Είχαμε συμφωνήσει, ε, ενώ δεν ήσασταν παρόν, ότι θα περάσουμε στη γνωμοδότησή σας. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να μην προβώ σε αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης που εκπώνησα, αλλά θα ήθελα να επισημάνω μόνο ορισμένα σημεία τα οποία πιστεύω ότι χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή μας. Το πρώτο αφορά το μέγεθος του προπολογισμού. Λαμβάνοντα υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου και τι εξελίξει των διαπραγματεύσεων για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, Όλοι γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε μια αισθητή μείωση στα επίπεδα του προπολογισμού. Για το 2014 οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Για την πολιτική συνοχή η πρόταση της Επιτροπής συνιστά μείωση 13,5% στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 9,3% στις πληρωμές. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή το 52% των πληρωμών για το 2014 πρόκειται να διατεθεί για την πληρωμή εκκρεμών λογαριασμών από προηγούμενα έτη, αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό καθώς τα ράλς συνεχίζονται να αυξάνονται. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού στηρίζει τις συνολικέ της εκτιμήσει, στην υπόθεση ότι τα επιπλέον 11,2 δις ευρώ στις πληρωμές που έχει ζητήσει μέσω του σχεδίου διορθωτικού προπολογισμού του 2013 θα έχουν πλήρω εγκριθεί κατά τη διάρκεια του έτου αυτού. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σα και θεωρώ ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Επιτροπή μα αφορά το γεγονό ότι η Επιτροπή έλαβε ω βάση για το ποσοστό προχρηματοδότηση στη θέση του Συμβουλίου. Ωστόσο αυτό είναι ένα ζήτημα που αποτελεί μέρο των συνεχιζόμενων τρεμερών διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό των κοινών διατάξεων, το γνωστό CPR Regulation, και πρόκειται στη διαδικασία της, υπόκειται στη διαδικασία της συναπόφασης. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε η Επιτροπή να προκαταλάβει με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους κατά την έναρξη της περίοδου να πληρώσουν εκ των προτέρων χρήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η επένδυση στα έργα που θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τρίτον, αναφορικά με την αύξηση των ποσοστών στη χρηματοδότηση co-financing rates top-up και τη χαλάρωση των κανόνων αποδέσμευσης the commitment rules για ορισμένα κράτη-μέλη, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας ενημερώσει η Επιτροπή εάν έχει υπολογίσει το πιθανό αντίκτυπο των δύο προτάσεων στον προπολογισμό του 2014. Με αυτή την ερώτηση βάζω μια τελεία στην παρέμβασή μου και αναμένω να πάνε της Επιτροπής καθώς και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς από την Επιτροπή που θα ήθελε το λόγο. Όχι. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Όχι. The deadline for amendments. Προθεσμία για τροπολογίες μέχρι τις 18 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Οπότε, περνάμε στο επόμενο θέμα. 15. Ευρωπαϊκό εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013. Παρακαλώ τον εισηγητή, κύριο Τάμας Τόιτς, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συνάδελφε. Το σχέδιο γνωμοδότησής μου βασίζεται σε δύο προηγούμενα κείμενα που συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα πρέπει να έχετε υπόψη και αυτά τα δύο προηγούμενα κείμενα, μια έκθεση και μια γνωμοδότηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μερικά ε, ζητήματα που αφορούν το θέμα αυτό για να ξεκινήσουμε την ουσιώδη συζήτηση από αυτού. Πρώτα απ' όλα, δημιουργία θέσεων εργασία. Η σημασία τη δημιουργία θέσεων εργασία είναι πολύ βασικό ε, σημείο του κειμένου μου. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει κανείς να υποτιμήσει τη σημασία αυτού του σημείου. Είναι το πιο σημαντικό. Η πολιτική συνοχή πρέπει να έχει τι αναγκαίε πιστώσει, στη διάθεσή της για να υπάρξουν οι κατάλληλες επενδύσεις και τονίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι οι κύριοι λήπτες ε, επενδύσεων μέσω των προσπαθειών μας. Ξέρουμε ότι σε όλες τις χώρες της Ένωσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι και οι σταθερότερες. Γι' αυτό η πολιτική συνοχής μας πρέπει να έχει την αναγκαία χρηματοδότηση είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και ακόμη περισσότερο να αναφερθώ στην ε, ε, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Τώρα έχει προαναφερθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση με την οποία συμφωνώ. Είμαστε φυσικά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αυτό δημιουργεί ανησυχίες και ένα περιβάλλον στο οποίο οι επενδυτές ε, ε, διστάζουν να επενδύσουν, αναβάλουν τις επενδύσεις τους και αυτό έχει αρνητική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές για επενδύσεις. Να τους καθισχάσουμε, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανάληψη κινδύνων. Δηλαδή ένα σταθερό και αποτελεσματικό διοικητικό πλαίσιο, να μειωθεί η γραφειοκρατία και βεβαίως να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Τώρα να περάσω στην μακροοικονομική διακυβέρνηση. Αναφέρω στην γνωμοδότησή μου και το θέμα αυτό. Καλωσορίζω το ότι στο τέλος Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε την κατάσταση σε διάφορα κράτη-μέλη και αποφάσισε ότι θα πρέπει να σταματήσει η διαδικασία υπερβολικού ε, ελλείμματος. Ε, αυτό αποφασίστηκε συγκεκριμένα και για την Ουγγαρία και είναι βέβαια θετικό από, από πλευράς μακροοικονομικής διακυβέρνησης. Και καταλήγοντας, Πρόεδρε, τονίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην καταπολέμηση της ε, απασχόλησης, στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επενδύσεις, στην εξυγίανση της οικονομίας μας, βιώσιμες επενδύσεις και φυσικά σε όλα αυτά οι πόροι της πολιτικής συνοχής παίζουν μεγάλο ρόλο και γι' αυτό οι πόροι της πολιτικής συνοχής πρέπει να είναι επαρκείς ιδιαίτερα λοιπόν μέσω των διαθροτικών ταμείων και την Τράπεζα μερίσων. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόιτς. Η κυρία Κλέβα. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης, διότι πραγματικά είναι πολύ καλή η διάρθρωση. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κοιτάζουμε πραγματικά όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και είναι πολύ καλός τρόπος να δούμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από το πρίσμα της περιφερειακής πολιτικής έτσι όπως το παρουσιάζεται. Ένα από τα βασικά θέματα του Ευρωπαϊκού Εξαμεινού είναι ο κύκλος, δηλαδή παρόμοια έγγραφα που υποβάλλονται ετησίω αλλά ζωτική σημασία εφόσον του δώσουμε την κατάλληλη προσοχή ώστε το Κοινοβούλιο να ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίες συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δίνουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις, αλλά συνολικά δεν έχουν πείσει ω προς την ε, ισορροπία και το εύστοχο των πολιτικών στόχων αναπολιτικό τομέα. Η κρίση δεν έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε έναν ε, κοινό τρόπο ε, να προχωρήσουμε, κάτι που ίσως να είναι άπιαστο όνειρο. Ε, πάντως, οι τομείς στους οποίους δίνεται προτεραιότητα και έμφαση στην έκθεση αυτή, ανα, ανάπτυξη, ανεργία, ε, και πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι πολύ καλά επιλεγμένες. Ο εισηγητής σωστά ε, επισημαίνει την ε, συνεχή μείωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και το πώς χρειάζεται ενίσχυση από τα διευθυντικά ταμεία στην τόνωση, για την τόνωση των επενδύσεων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, η έλλειψη επενδυτικών ικανοτήτων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανησυχία μου γι' αυτό θα πρέπει να διασυνδεθούν με το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίω στι λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ. Εκεί δεν βλέπουμε να επιτελείται πρόοδο μεταξύ ε, ε, για την ανάκτηση λόγου χάρη των δυνατοτήτων των τραπεζών και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων. Ω προ την ε, ανάκτηση πόρων, νομίζω ότι το ε, δημοσιονομικό εργαλείο θα μπορούσε να είναι ένα από τα μέσα που θα μπορούσαμε, από τα από τα μέσα θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στην πολιτική συνοχή. Τα διευθυντικά ταμεία έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, όπω επισημαίνει και ο εισηγητή στην παρουσίασή του. Και τέλο, καλώ ε, επικεντρώνεται ο εισηγητή ε, στην ανεργία και μάλιστα την ανεργία των νέων για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα μπορεί να διαδραματίσει εδώ και ένα ρόλο και η πολιτική συνοχή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά αυτά υπόψη στα πλαίσια των διπλωματεύσεων για το πακέτο της συνοχής αλλά και το τι θα γίνει με τα διευθυντικά ταμεία. Το καλωσορίζω λοιπόν την τοποθέτηση του συγγητή και τις προτάσεις του και για το θέμα αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Κλέβα. Κάποια άλλη ερώτηση παρέμβαση ο κύριος Ρόι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για τον αντίκτυπο το τι γίνεται με τα υπόλοιπα προς ακαθάριση. Τα ραλ της πολιτικής συνοχής για το 2013. Πώς θα επηρεαστούν οι οι δαπάνες της επόμενης χρονιάς, οι ικανότητες για δηλαδή, δαπάνες. Πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα. Δεν θα μεταφερθούν πολλοί λογαριασμοί για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Πώς ε, θα επηρεάσει αυτό. Μπορείτε να μας δώσετε τον αριθμό. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Φανίστερ Κύριε Ντόιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που μας εξέφρασαν τις απόψεις τους. Νομίζω στην ερώτηση του κυρίου Φανιστεροή καλύτερα να απαντήσουν οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως βρίσκονται εδώ ε, στην αίθουσα. Ίσως αν τους δώσετε το λόγο κύριε Πρόεδρε να μπορέσουν να δώσουν και τα αριθμητικά στοιχεία για το θέμα για το θέμα του που έθεσε ο κύριος Φανίσταροι Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμφώνησαν με, το, με τα βασικά στοιχεία της ε, γνωμοδότησης, αλλά νομίζω ότι γενικά υπάρχει ευρία συνένεση παρά τις τροπολογίες που μπορεί να υποκληθούν. Ευχαριστώ κύριε Σιγητή, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα φροντίσω να τους σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα. Με αυτά θα ήθελα να διακόψω τη συνεδρίαση ως τις 11. Αν με συγχωρείτε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. So, as I όπως σας είπα, διακόπτουμε ως τις 11. Ευχαριστώ.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

Είναι μια μορφή που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να χρησιμοποιήσω τα πλήρια του. Επίση, είναι μια μορφή που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να δημιουργήσω τα να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 Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ως συνήθω θα κάνουμε μια ψηφοφορία ελέγχου. Παρακαλώ, βάλτε την κάρτα σας να ελέγξουμε εάν λειτουργούν όλων οι κάρτες. Άρχεται. I understand that people who are here... Uh, μου φαίνεται ότι... Α, ωραία, έληξα. Δεν έχει κανείς πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, αρχίσουμε το γενικό κανονισμό. Παρακαλώ, υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, βάλτε πάλι τις κάρτες σας ε, στο μηχάνημα. Ωραία. Block vote, ψηφοφορία ε, κατά τμήμα υπέρ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνολική ψηφοφορία 2, υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 27 στη σελίδα 4. Τροπολογία 27. Στη σελίδα 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 951. Σελίδα 9. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 σελίδα 11 Υπέρ λοιπόν 56 λέει τώρα κατά αποχές εγκρίνεται σελίδα 12 τροπολογία 67 Σελίδα 12, 67 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 στην επόμενη σελίδα. Σελίδα 13 τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 20 τροπολογία 119. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, να ελέγξουμε. Την τροπολογία 119. Mm. Άρχεται. Ψηφίζει ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Πρέπει ένας να βγάλει την κάρτα του παρακαλώ. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Εντάξει, ωραία. Πέρας εγκρίνεται. Ε, γιατί έπρεπε να ελέγξουμε δηλαδή. 40 με 4. 179 σελίδα 26. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 29. 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στη σελίδα 30 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην επόμενη σελίδα 493. Ήταν στην ψηφοφορία σε μπλοκ. Σελίδα 31. 493 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 38. 282 σελίδα 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 284 λίγο παρακάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σελίδα 43 499 σελίδα 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σελίδα 44. 3, 4, 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 46. 355. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 σελίδα τώρα 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 από κάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σελίδα 55 έχουμε τις γνωμοδοτήσεις έχουμε την ψηφοφορία σε μπλοκ 3 σελίδα 55 για τις νομοδοτήσεις παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σελίδα 56 έμπλ 14 για την αιτιολογική σκέψη 57 57α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά 64, 148, συγγνώμη, έμπλα. Σελίδα 64, τροπολογία 148, έμπλα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Α, ναι, ναι, βεβαίως. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην απέναντι σελίδα. 153 έμπλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 έμπλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σελίδα 70 έμπλ 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην επόμενη σελίδα 230 έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία δεν το πιστεύω ηλεκτρονική παρακαλώ άρχεται Ψηφίζουμε την νομοθετική τροποποιημένη πρόταση. Άρχεται. Πέρας. Ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα νομοθετική πρόταση. Θα, λήξει. Αν δεν θέλετε να ψηφίσετε, μην ψηφίσετε. Πέρασε. Και έχουμε 40 υπέρ 3 κατά μία αποχή. Σιγά περιμένετε το την νομοθετική πρόταση. Καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι ακόμη η νομοθετική πρόταση. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε και το νομοθετικό ψήφισμα, ηλεκτρονικός και πάλι, άρχεται. Yes, 41 υπέρ, 3 κατά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να ψηφίσουμε και κάτι ακόμη, αλλά ε, διανατάσεως. Μπορεί να προκύψει η κατάσταση όπου θα χρειαστεί να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μας δώσετε την εντολή για να ξανα αρχίσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την εντολή και με βάση την έκθεση που μόλις εγκρίναμε με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Σας παρακαλώ λοιπόν να χορηγήσετε στην διαπραγματευτική μας ομάδα αυτή την εντολή. Παρακαλώ ποιοι είναι υπέρ αυτών που είπα. Κατά αποχές. Ωραία, χορηγήσαμε και αυτή την εντολή. Και συγχαίρω την Κωνσταντσε, τον Λαμπέρ. Ξέρω ότι ίσως θα να πούν δύο λόγια να ξεκινήσει ο Λαμπέρ. Μία πρόταση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία για ένα τόσο περίπλοκο θέμα και ιδιαίτερα για την καλή του θέληση συνεργασίας που μας επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι μιλώ και εκ μέρους της Κωνσταντσε και όλων των σκιωδών ευχαριστώ. Νομίζω και η Κωνσταντσε θέλει να τα πει, όχι. Αν δεν θέλει να μιλήσει. Συμφωνώ απόλυτα με τον ε, Λάμπερτ. Όλα πήγαν άψογα και ευχαριστώ τους πάντες. Αλλά δεν ήταν πάντα τόσο καλά τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πει τίποτα. Ωραία. Να περάσουμε στο Περιφερειακό Ταμείο που είναι το επόμενο θέμα. Τροπολογία 29. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Κατά τμήματα. Τρία τμήματα. Να αρχίσουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές ευχαριστώ ε, το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να την 96 άρχεται εγκρίνεται 36 τώρα, όχι όχι 34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 κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ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 Περνάμε τώρα στις γνωμοδοτήσεις. Η Κωνσταντς. Μία ερώτηση, ίσως έκανα λάθος, αλλά γιατί δεν ψηφίσαμε την 67. Η 67 στη σελίδα 6. Δεν την ψηφίσαμε. Α, πρέπει να την ψηφίσουμε. Κωνσταντζε, ακόμη και ο Όλμπριχτ ε, δεν ξέρει που βρίσκεται, αλλά χωρίς εσένα, όχι μόνο ο Λαμέρλα και ο Γιάννη. 67, πρέπει να ψηφίσουμε. Σελίδα 6. 67 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Περνάμε στις νομοδοτήσεις. Uh, uh, Τώρα θα ψηφίσουμε on block τις ε, τροπολογίες που έχουν καταπέσει. τις τροπολογίες που δεν έχουν καταπέσει. Ωραία. Ομαδικά. Συμφωνείτε, καταλαβαίνετε τι ψηφίζουμε. Εφόσον το καταλάβατε, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ίδιο για την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας και ασφάλεια συντροφίμων. Οι τροπολογίε που δεν έχουν καταπέσει θα ψηφιστούν ομαδικά. Πού είναι. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Σελίδα 13. Ήτρε. Βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Οι τροπολογίε που δεν έχουν καταπέσει ψηφίζονται ομαδικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Και τώρα στη σελίδα 18. Μεταφορές και τουρισμός. Το ίδιο. Τροπολογίες που δεν έχουν καταπέσει ψηφίζονται ομαδικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Εάν έχετε κάτι να πείτε, πείτε το τώρα. Δεν υπάρχουν σχόλια. Ωραία. Περιμένουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Παρακαλώ. Βάσει των όσων σημείωσα, δεν ψηφίσαμε την 68 και 69. Την 67 την περάσαμε. Αλλά έχουμε και την 68 και 69. Δεν ψηφίστηκαν και κοίταζα τώρα. Έκανα έλεγχο με τον κατάλογο. Εδώ δεν έχει σημειωθεί ότι πρέπει να ψηφιστούν στη σελίδα 6 στο δικό μου κείμενο, μετά την 67. Εσείς λέτε και για την 68 και την 69 ότι πρέπει να ψηφιστούν και αυτές. 68 λοιπόν, υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται και 69. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω αν χρειαστεί αλλά πρέπει να κάνουμε και την τελική ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 για 4 εποχές. Εντάξει, και το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνατε με δύο εποχέ. Τελειώσαμε και με αυτό. Συγχαρητήρια στον κύριο Όλμπριχτ. Για αν κάποιος ήταν υπεράριθμο, μια ψήφο παραπάνω υπέρ. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με τους σοσιαλιστές. Εντάξει Γιάννη, έχεις το λόγο. Απλώς να πω ότι δεν ήταν καθόλου απλές οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι μακροσκελής ο κανονισμός, αλλά απέτησε μια στάση ιδιαίτερα διαλλακτική και ανοιχτή από την πλευρά της διαπραγματευτικής ομάδας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την κοινή μας δουλειά. Κάποιες φορές δεν συμφωνούσαμε, αλλά η τελική ψηφοφορία δείχνει ότι τελικά έχουμε κάποια κοινή συνεννόηση για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Όντω, τα πράγματα κάποιε φορέ ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Αλλά χάρη στην παρέμβαση του Γιάννη και άλλε μεταπτυχιακέ ομάδε τα καταφέραμε. Για αυτή την ψηφοφορία πρέπει να πω ότι σα ζητάμε ταυτόχρονα και την ε, εντολή, την διπλωματευτική εντολή σε περίπτωση που χρειαστεί να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Ε, συμφωνείτε να συνεχιστεί η διαπραγματευτική εντολή. Ε, Αντιρρήσει, αποχέ, ωραία. Κλείσαμε και με αυτό. Περνάμε στον Βίκτορ. Ταμείο συνοχή.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση προπολογισμών. Τροπολογίε Επιτροπή Προπολογισμών. Ό,τι δεν έχει καταπέσει ψηφίζουμε ομαδικά. Unblock. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτονται. Envy. Το ίδιο. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτονται. Ήτρε. Υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτονται. Τραν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία. Σε δύο σκέλη. Η νομοθετική πρόταση ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Μπορούσα να το κάνω και μόνη μου. Δεν ήταν ευγενικό όμω. Με συγχωρείτε. Δεν έχω τον κατάλογο και ξέχασα κάποιον που Λοιπόν, 45 μία εποχή. Βίκτορ. Ήταν νικηφόρος η έκβαση. Για, τη δεύτερη, για το δεύτερο σκέλος, νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. 43, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Τελειώσαμε. Θες να πεις κάτι? Ε, συγκίνηση. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστίες ε, στους ε, εξαιρετικούς σκιώδεις εξηγητές όλων των πολιτικών ομάδων. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Ήταν αξιοσημείωτη η εμπειρία αυτή για τη ζωή ενός ανθρώπου να έχει συνεργαστεί κατά αυτόν τον τρόπο με τόσο διαφορετικούς ανθρώπους από τόσο διαφορετικές προελεύσεις και με τέτοιο διαφορετικό ιστορικό. Αλλά φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα σύμπνοιας. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Πίτερ Μπέρκ για την διάρκεια του στήριξη και Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τους διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και προσώπους συλλόγων και ε, βιομηχανικών ε, ενώσεων, διότι μας στήριξαν και πετύχαμε κάτι έξω σημείο. Τον έχουμε τις ίδιες διατάξεις για δύο ταμεία, τα οποία είναι θεμελιώδη σημασία για, την... για τι κοινότητέ μα. Ευχαριστώ και την Κάρλα από την Γραμματεία και τον Τάριο για την ε, φοβερή δουλειά που έκαναν μας βοήθησαν πάρα πολύ και είναι ένα πολύ καλό νομοθέτημα αυτό. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Ευχαριστώ. Θέλω την έγκρισή σας παρόλα αυτά. Διαπραγματευτική εντολή για τον Βίκτορ σε περίπτωση που προκύψουν εξελίξεις που θα απαιτήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωρούμε, η Δυστυχώς ο Ρίκα Μάνερ δεν είναι μαζί μας, αλλά έχει κάνει φοβερή δουλειά. Ελπίζω να είναι και η ψηφοφορία μας παρόμοια. 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται.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 Συμβαστική 2 υπέρ. Όχι. 56, συγγνώμη. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά υπέρ είναι κανείς υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται, 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 3 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ θα μπορούσα να τον μπλοκάρω να τα ψηφίσουμε όλα μαζί ίσως μπορούμε να τις ψηφίσουμε δεκά. από 25 ως 100 το δέχεστε μέχρι τις νομοδοτήσεις, μέχρι τα 38 να ψηφίσουμε αυτή τη σελίδα μαζί όλες τις τοπολογίες. Ωραία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Από το 24 ως το 38, δηλαδή μέχρι τις νομοδοτήσεις, εγκρίνονται. Νομοδοτήσεις τώρα. Πρώτα απ' όλα, μπουτ, Το προπολογισμό. Το ίδιο. Όσε δεν έχουν καταπέσει, ψηφίζονται οντοματικά υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ε, κοντ, το ίδιο σύστημα υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τραν, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και τελειώσαμε. Τελική ψηφοφορία. Δύο τελικές ψηφοφορίες. Νομοθετική πρόταση όσο τοποποιήθηκε. Θέλεις να πεις κάτι Κωνσταντ. Όχι. Απλώς βγήκες. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πολύ ωραία. 43. Μία ψήφος κατά δύο εποχές. Νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 42-1-2. Τέλεια. Δεν είναι εδώ η Ρίκα, αλλά σίγουρα θα είχε κάτι να πει. Μόλις γέννησε, όπως ξέρετε, έκανα αγοράκι αλλά μου τηλεφωνάει και με ρωτάει πώς ε, προχωράνε τα πράγματα. Ενδιαφέρεται δηλαδή ακόμα για τις υποθέσεις μας. Οπότε και εκ μέρου της σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συμβάλλατε στην επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Τώρα, διαπραγματευτική εντολή για ό,τι επίγον προκύψει. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, Υπάρχει πρόταση από τον κύριο Τσέλερ που ήταν πολύ καλός διαπραγματευτής. Νομίζω ότι τα κατάφερε σε όλα. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί, ομαδοποιημένα όλες του τις τροπολογίες, αν συμφωνείτε. Ποιοι είναι υπέρ όλων των τροπολογιών λοιπόν που προτείνει ο Γιακίμ Τσέλερ στον κανονισμό αυτό για τον όμιλο δαφικής Κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα περνάμε στις δύο τελικές ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα για την τροποποιημένη νομοθετική πρόταση. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 42 υπέρ, 3 αποχές. Νομοθετικό ψήφισμα τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Πάλι το αποτέλεσμα 40 υπέρ, 2 αποχές. Συγχαρητήρια Ιωακήμ. Διαπραγματευτική εντολή τώρα. μήπως χρειαστεί. Χρειαστούν κάποιες προσαρμογές, υπάρξει κάποιο σφάλμα. <clears throat> Λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται για πραγματευτική εντολή. <clears throat> Ιωκίμ, έχεις κάτι να πεις? Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, Ευχαριστώ για την ε, έγκριση του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να ευχαριστήσω την πρόεδρό μας, κυρία Χίμπνερ, η οποία συμμετείχε, μας υποστήριξε. Εσείς καταφέρατε να προχωρήσει το θέμα αυτό σε αυτή την περίοδο και αυτά που κάνουμε τώρα είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για την ε, διαμεθοριακή συνεργασία. Και τώρα θέλουμε να διαβρύνουμε τις δυνατότητές του. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία της ε, Επιτροπής και κυρίως τον κύριο Μάνεφ που μας υποστήριξε, τον βοηθό μου, τον σύμβουλο δόκτωρα Κάλιτα από την ομάδα μου και βεβαίως ο βοηθός μου ε, συμμετείχε ιδιαίτερα, ανέλαβε το κύριο βάρος τον οργανωτικών προσπάθειων. Ευχαριστώ και την Ιρλανδική Προεδρία που συνέβαλε πολύ για τις διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν απλό αυτό. Δεν ήταν απλό να αντιμετωπίσει ε, και να παρουσιάσει μια θέση του Συμβουλίου με την οποία πολλοί δεν συμφωνούν και ορισμένοι, δηλαδή ορισμένα κράτη-μέλη, δεν το γνωρίζουν καν αυτό το νομικό μέσο. Οπότε οι διαπραγματεύσεις ορισμένες φορές οδήγησαν σε συγκινήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επιτροπή, τον κύριο Πέτερς, ο οποίος ήταν πάντα στο πλευρό μας και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επιτροπή Περιφερειών. Αυτό είναι το μέσο εργασίας για την διαμεθοριακή συνεργασία περιφερειών. Ήδη έχουν δημιουργηθεί 30 περίπου τέτοιες ε, δυνατότητες εδαφικής συνεργασίας, ευρωπαϊκή όμιλη εδαφικής συνεργασίας και αυτοί μας επιτρέπουν όχι μόνο να εργαστούμε ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις όμορες χώρες. Πρέπει λοιπόν πολλούς να ευχαριστήσω και ευχαριστώ και εσάς για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και για τις διαπραγματεύσεις που περαιτέρω πρέπει να διεξαγάγω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, σε 45 λεπτά έχουμε προχωρήσει. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Κλέβα. Πρόκειται για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Μια στιγμή. Δεν θα λέγω ότι κοιμάμαι, ίσως όμως έχω κουραστεί. Υπάρχουν τρία τμήματα στη συμβαστική. Ένα πρώτο τμήμα υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα, γιατί έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία, τη συμβαστική αριθμό 1. Πρώτο τμήμα λοιπόν, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε πριν κλείσουμε την ψηφοφορία, πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Πάλι θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε επίσης. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα. είναι περίπλοκο. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 26 εξαιτία της περίεργη κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε. Υπέρ λοιπόν, τροπολογία 26. Κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 26. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίες. Απορρίφθηκε. 28 τώρα, τροπολογία 28. Υπέρ. Α, θα ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι είναι η ίδια πλειοψηφία, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε λοιπόν για την τροπολογία 28. Πέρα τη προφορία. Απορρίφθηκε επίσης με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 3. Υπέρ. Α, έχει δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Μια που έχουμε χρόνο, ας ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα συμβαστικής 3. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ίδια πλειοψηφία όπως και πριν. 25 κατά 19 υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 τώρα. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Τροπολογία 35. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της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 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές α θα ελέγξουμε για την 61 ψηφίστε παρακαλώ τροπολογία 61 πέρα στις ψηφοφορίες 22-22 απορρίπτεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ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 Εγκρίθηκε 23 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Η 76 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 79. Ψηφίστε παρακαλώ. Λαμπέρ. Δεν έχω τον κατάλογο ψηφοφορία σας, γι' αυτό σας κοιτάω. Έχω ένα πρόσχημα έτσι για να σε κοιτάω, Λαμπέρ. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία Εγκρίθηκε. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 82, ψηφίστε. Πέρα τη εγκριθηκε Εγκρίθηκε. 22-21. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Α, 89 θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Α, όχι, θα ελέγξουμε για την 90. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 90. 2 καταπίπτει. Σωστά. όχι. 92. Ψηφίζουμε το 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93. Είναι κανείς κατά της προφορικής. Όχι, έτσι. Ωραία. Τι τροποποιημένη τροπολογία λοιπόν. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά Καλά, σε ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίες απορρίφθηκε. 20-24 ε, κατά. 100 την ψηφίζουμε. Ναι, 100, τροπολογία 100. Πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε την 99. Τροπολογία 99 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 100. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά απορρίπτεται νομίζω αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 104 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορίας απορριφθήκε 18-25. 105 υπέρ κατά θα ελέγξουμε για την 105 ψηφίστε. Όχι ακόμα. Περιμένετε. Τώρα. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίφθηκε με 27 ψήφους κατά 18 υπέρ, 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ, κατά, δεν ξέρω, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, 110 ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 27 κατά, 18 υπέρ. 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Θα ελέγξουμε και για την 107 γιατί δεν είμαι σίγουρη. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 100... Πού είμαστε τώρα? 108. Ψηφίζουμε το 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 119, α δεν την ψηφίσουμε. 121 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Θα ελέγξουμε. 129 ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Απορρίφθηκε. 25 κατά, 19 υπέρ. 130 τώρα, σωστά. Υπέρ. 130 υπέρ. Έχω υπομονή. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135. Έχει, υπάρχει και τροποποίηση, είναι κανείς κατά. Όχι, ωραία. Την τροποποίηση τροπολογία λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Θα ελέγξουμε για την 136 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 24 ψηφικά κατά, 21 υπέρ. 137 τώρα υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 137. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 25-20. 138 υπέρ. Πάλι θα ελέγξουμε. 138 ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίστε. Πάλι το ίδιο 25-18 απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Εδώ έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, θα ελέγξουμε για την 147. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. <clears throat> Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε 25 κατά 20 υπέρ, 148 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά θα ελέγξουμε. 149. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίφθηκε 24 κατά 19 υπέρ, 150 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 151 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 152 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 153 υπέρ. Θα ελέγξουμε για την 153. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 24 κατά 21 υπέρ. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροφολογία 1 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές συγκρίνεται 14 υπέρ, θα ελέγξουμε για την 104, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. <clears throat> Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε 25 κατά, 20 υπέρ, 15 τώρα υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για την 15 επίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορία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 Ηλεκτρονικά λοιπόν, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 20 κατά ήτρε 3 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Φαντάζομαι ίδια πλειοψηφία, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε 5. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορία. Εγκρίνεται 25 υπέρ, 20 κατά. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. 9. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 20 κατά 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε τι άλλε που έχουν καλυφθεί. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, έτσι. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 37 υπέρ, 2 κατά, 6 αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια. Περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα, επόμενη ψηφοφορία. Πού είναι η έκθεση της Εμίλια Ματσόνη δημοσιονομικοί περιορισμοί για, τις, ε, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 προφορική. Έχει καμί... κανείς αντίρρηση. Όχι. Ωραία. Τροπολογία 18 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 23 υπέρ. Να ελέγξουμε την 23. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ 24 ε, κατά. Για την 3 υπάρχει προφορική, είναι κανείς κατά, όχι, ωραία, ψηφίζουμε. Την τροποποιημένη συμβαστική 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, συμβαστική 4. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται ψηφίζουμε τη 49 με προφορική τροπολόγηση ψηφίζουμε λοιπόν 49 να ελέγξουμε τη 49 όπως τροποποιήθηκε άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ 17 κατά. 47 υπέρ. 47 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αν θέλετε να ελέγξουμε, ωραία, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 47. Πέρασε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 Παρακαλώ μην μιλάτε γιατί μετά δεν ψηφίζετε και χάνετε. Και εγκρίνεται 28 υπέρ 16 κατά. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. 7 λέγω. Οι σοσιαλιστές δεν ξέρουν οπότε Λαμπέρ ε, μπορεί και να περάσει. Λοιπόν, 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 με την προφορική τροπολόγηση δεν υπάρχει αντίρρηση ωραία ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται προτάσεις ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ 5 υπέρ Ωραία, να ελέγξουμε την πρόταση, την σύσταση 5 των προϋπολογισμών. Πέρας. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Να ελέγξουμε και την 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, απασχόληση 1. Ένα έμπλα. Ε, υπέρ απορρίπτεται. 4. Είναι όλε ε, ε, συμβαστές. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλε μαζί. Μία έω 11. Α, όχι. Καλά, εντάξει, ωραία. Ωραία, είμαστε στην 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Α, ναι, πρέπει να ελέγξουμε την 5.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 Πέρας. Και εγκρίνεται. 23 με 22. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12, όχι εντάξει, 15 υπέρ. Να ελέγξουμε τη 15. Άρχεται. The closed. Πέρας. Εγκρίνεται 23 με 22. Α, και η τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. 40 υπέρ 2 κατά. Μία πρόταση παρακαλώ, Ερμηνεία. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή, ευχαριστώ τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτό η Επιτροπή Ρέτζη και το Ευρωκοινοβούλιο έδειξε ότι πραγματικά έχει ξεπεράσει τις ε, εθνικές και ευρωπαϊκές γραφειοκρατίες ξεκινά ένα σύστημα που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κατευθυνθεί προς μια αυστηρή πολιτική μεν, αλλά και ανάκαμψης. Διότι ιδάλλως θα εγκρίναμε μια αντιευρωπαϊστική πολιτική. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στη Μαρία Ιριγκόγεν Πέρες για την επαναβιομηχανοποίηση. Τροπολογία 1. Να περιμένουμε λίγο γιατί το ΕΛΚ δεν ξέρει να ψηφίζει. 1. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά τμήματα χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχή. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολόγια 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 με προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία, όχι. Οπότε ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 8. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 9. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, έληξη ψηφοφορία. 42, τρεις αποχέ. Εγκρίνεται, συγχαρητήρια Μαρία. Uh, yes, Mr. Λαμπέρτ, κύριε Φανίστερο, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερω εσάς για αυτή την τόσο αποτελεσματική διεξαγωγή της ψηφοφορία για όλα αυτά τα πακέτα. μας φέρατε σε αυτό το θετικό πέρας και πολλές ευχαριστίες και στη γραμματεία της Επιτροπής μας. Πραγματικά ήταν μεγαλειώδες το έργο σας. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, θέλατε να μας πείτε ότι τα πήγαμε καλά. Στα Ολλανδικά μπορεί να τα λέγατε διαφορετικά, να επικρίνατε. If we can have this afternoon after the, the, the uh, dear colleagues. Συνάδελφοι, επειδή είναι ακόμη εδώ ο κύριος Βίνκλερ και το δικό του σημαίνει το τελευταίο αύριο στην ημερήσια διάταξη και μετά τη Λιθουανική Προεδρία ίσως να μην χρειαστεί να συνεχίσουμε ε, αλλάζουμε ίσως τη σειρά και κύριε Βίνκλερ αν θέλετε μπορείτε να παρουσιάσετε τώρα την εκθεσή σας. Θα έχουμε λοιπόν στις 3 την έκθεση Βίνκλερ.